Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Αρχίζουμε ευθύ αμέσω τη συνεδρίασή μας. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ήρθατε στην απογευματινή μας συνεδρίαση που αρχίζει με ένα πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και αυτό εν ώψη της επερχόμενης ε, επίσκεψης που θα κάνουμε στην Ιαπωνία. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν, και θεωρώ ότι είναι προνόμιο για μένα που μπορώ να υποδεχτώ εδώ την εξοχότητά του, τον κύριο Καζούο Κοντάμα, που είναι ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλωσορίζω επίσης την κυρία Τερέζα Φαλών η οποία είναι ε, ξέχουσα ερευνήτρια, αλλά και πολύ γνωστή δημοσιογράφος και σύμβουλος για πολλά θέματα ασφάλειας. Οπότε, κύριε Πρέσβη, ε, κυρία, καλώς ήρθατε στην ε, συνεδρίαση αυτή της Υποπιτροπής Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το σημερινό μας θέμα, λοιπόν, είναι η πολιτική ασφάλειας και άμυνας της Ιαπωνίας και σχετικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην πολιτική αυτή πρόσφατα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ασφάλειας. Στη συνέχεια έχουμε δημόσια κρόαση, οπότε δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Θα δώσω το λόγο ευθύς αμέσως στην εξοχότητά του τον πρέσβη της Ιαπωνίας και μετά στην κυρία Φαλών. Παρακαλώ. Έφτασε και ο τρίτος προσκεκλημένος μας. Οπότε να σας τον παρουσιάσω, αν και τον γνωρίζετε ήδη πιστεύω. Είναι ο διευθυντής Γκούναρ Βίγκαντ. Είναι διαχειριστικός διευθυντής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης όσον αφορά την Ασία και τον Ειρηνικό. Είναι ο τρίτος μας μιλητή σήμερα για να συζητήσουμε και μαζί του τα θέματα της παγκόσμιας ασφάλειας και πιο συγκεκριμένα τη συνεισφορά της Ιαπωνίας σε αυτήν. Να δούμε δηλαδή πώς η Ιαπωνία συμμετέχει στην διεθνή σκηνή ασφάλειας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, εξοχώτης. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Υποβιτροπής αυτής Ασφάλειας και Άμυνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρία Φωτίγκα αξιότιμοι ευρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής αυτής, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι μεγάλη τιμή για μένα και χαρά που προσκλήθηκα σήμερα στην Επιτροπή σας. Από την προηγούμενη χρονιά η πριγκίπισσα Τικάμι προσκλήθηκε να έρθει και να μιλήσει στην Επιτροπή αυτή για να εξηγήσει τι εννοούμε όταν μιλούμε για την συνεισφορά της Ιαπωνίας στην ειρήνη, επικεντρωνόμενη κυρίως στο γεγονός ότι η Ιαπωνία σκόπευε να αναθεωρήσει την νομική δομή που είχε να κάνει με τη διεθνή συνεργασία, την ασφάλεια, με τις δομές ειρήνευσης ανά τον κόσμο κλπ. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσω μετά από εκείνη την παρουσίαση την περσινή για να σας δώσω τις απόψεις της Ιαπωνίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις μας για την ασφάλεια και την άμυνα και ποιε πιστεύουμε ότι είναι υποπτώσεις στην σημερινή περιφερειακή ασφάλεια. Για να σας υπενθυμίσω λίγο. Κοιτάξτε τη σελίδα 1 που σας έχω δώσει που αναφέρεται στην ασφάλεια και την άμυνα. Με δύο λόγια. Η νέα νομοθεσία επιτρέπει στην Ιαπωνία να ανταποκριθεί ήπια σε οποιαδήποτε κατάσταση μπορεί να απειλεί την ειρήνη την ευημερία των ε, Ιαπώνων και να συνεισφέρει στην ειρήνη και τη σταθερότητα παγκοσμίω. Η Ιαπωνία θα συνεχίσει λοιπόν σε αυτό το δρόμο, μια που είναι ένας λαός που αγαπάει την ειρήνη, όπως έχουμε κάνει και όλα αυτά τα χρόνια από τότε που έληξε ο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είμαστε βασικός παράγοντας στη διεθνή κοινότητα και γι' αυτό θα συντονιστούμε με όλες τις ενδιαφέρομένε χώρες, χώρες, Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φροντίσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς την ειρήνη. Τώρα, θα αρχίσω με τη σημερινή κατάσταση ασφάλειας στην Ιαπωνία. 2017. Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί ιδιαίτερα εξαιτία των απειλών από την Βόρεια Κορέα, των πυρηνικών της και των βαλιστικών της δυνατοτήτων που μας έχουν φέρει σε μια νέα ανησυχητική κατάσταση. Οργάνωσαν 20 εκτοξεύσεις και δύο πυρηνικές δοκιμές πέρυσι, το 2016 δηλαδή μόνο. Πρόκειται για απειλή στη σταθερότητα στην περιοχή έχει προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει βία προκειμένου να επικυρώσει τις ε, διεκδικήσεις της, τις εδαφικές. Και όσον αφορά τον ανέριο χώρο και της Ιαπωνίας και τις γείτονες χώρες. Σελίδα 2. Τώρα, θα ήθελα να επικεντρωθούμε λίγο στην αυξανόμενη απειλή της Βόρειας Κορέας τους τελευταίους μήνες. Σελίδες 3 και 4. Η ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων και των πυρηνικών στην Βόρεια Κορέα, όπως σας είπα και νωρίτερα, μας έχουν φέρει σε ένα νέο επίπεδο απειλής. Τέσσερις βαλιστικούς πυράβλους ταυτόχρονα περίπου εκτόξευσαν και τρεις από αυτούς βρέθηκαν στην Ιαπωνική θάλασσα. Η ανάπτυξη λοιπόν των βαλιστικών ε, πυράβλων και τα πυρηνικά της Βόρειας Κορέας αποτελούν τεράστια απειλή. Θα δημιουργήσουν και νέες ανησυχίες γιατί πρόκειται για τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής και σχετικών τεχνολογιών. Όλα αυτά αποτελούν μεγάλη πρόκληση για την σταθερότητα παγκοσμίω. Θα πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε όλοι αποφασιστικά και να υποχρεώσουμε τη Βόρεια Κορέα να συμμορφωθεί με όλα τα ψεφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Εμείς παρακολουθούμε ιδιαίτερα προσεκτικά την κατάσταση και όσον αφορά τη δολοφονία του αδερφού του σημερινού ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Από ό,τι φαίνεται χρησιμοποιήθηκαν κάποιοι παράγοντες και πρόκειται για έγκλημα τελικά. Ένα έγκλημα το οποίο με τίποτα δεν μπορεί να ανεχθεί η Ιαπωνία. Η Βόρεια Κορέα έχει απάγει επίση σε πολλού Ιάπωνε πολίτε, ένα 13χρονο κορίτσι μεταξύ άλλων. Οι απαγωγέ αυτέ είναι ιδιαίτερα ανησυχητικέ υπονομεύουν την εθνική κυριαρχία της Ιαπωνίας και την ασφάλεια και τη ζωή των Ιαπώνων. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την κυβέρνησή μας. Χρειαζόμαστε συνεργασία. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ λίγο και στα θέματα που έχουν να κάνουν με την Νότια Κινέζικη θάλασσα, σελίδα 5 του εγγράφου που σας έχει διανεμηθεί. Η Ιαπωνία προσπαθεί να αποκαταστήσει τις τρεις αρχές όσον αφορά το δίκαιο της θάλασσας. Οι αρχές αυτές επιβεβαιώθηκαν και στην διάσκεψη που έλαβε χώρα πέρυσι και με την οποία συμφωνούν οι G7, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η βασική αρχή είναι ότι οι χώρες, τα κράτη, διευκρινίζουν τις διεκδικήσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου. Η δεύτερη αρχή είναι ότι οι κυρίαρχες χώρες δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν βία προκειμένου να προχωρήσουν στις διεκδικήσεις τους. Και η τρίτη αρχή είναι ότι τα κράτη προσπαθούν να διακανονίσουν τις διαφορές τους ειρηνικά. Όμως η Ιαπωνία ανησυχεί όλο ιδιαίτερος εξαιτία των αυξανόμενων περιπτώσεων που οδηγούν σε εντάσεις στη διεθνή κοινότητα. Τώρα, η νότια κινέζικη θάλασσα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία γιατί βρίσκεται ανάμεσα στην Ασία και την Ευρώπη και οι διενέξεις που υπάρχουν επ' αυτής ενδιαφέρουν ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και την Ιαπωνία και τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιαπωνία έχει υποστηρίξει το κράτος δικαίου στην θάλασσα αυτή και θα συνεχίσει η Ιαπωνία να συνεργάζεται με τις ενδιαφερόμενες χώρες και θα συνεχίσει να ζητάει τη συμμετοχή όλων των χωρών σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Νότια Κινέζικη θάλασσα και θα συνεχίσει τις προσπάθειές της για μια ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων βάσει του δικαίου της θάλασσας. Γι' αυτό και χαιρόμαστε για το διάλογο ανάμεσα στην ΑΣΕΑΝ και την Κίνα. Είναι ένας διάλογος ο οποίος πρέπει να γίνει βάση του διεθνούς δικαίου και βάση της αρχής της μη στρατιωτικοποίησης και της συγκράτησης στην περιοχή. Η Ιαπωνία πιστεύει ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα και η Ιαπωνία δεν θέλει μονομερείς αλλαγές του στάτους κουβό που θα οδηγήσουν σε εντάσεις. Τώρα πρέπει να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά που σας είπα, όμως ακριβώς γι' αυτό υπάρχουν πολλά ανησυχητικά φαινόμενα στην περιοχή και γι' αυτό η κυβέρνησή μας υιοθέτησε την ανοιχτή στρατηγική του ειρηνικού, σελίδες 6 και 7. Πρόκειται για μια ανοιχτή θάλασσα στον ειρηνικό υπέρ της ευημερία της διεθνούς κοινότητας. Η ενδορική περιοχή, δηλαδή η περιοχή στον ειρηνικό, περιλαμβάνει και κινέζικες και ινδικές περιοχές, όπως επίσης αφρικανικές περιοχές. Ο ειρηνικός λοιπόν είναι μια πάρα πολύ σημαντική θάλασσα. Πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτή τάξη στη θάλασσα αυτή, όπως προβλέπεται από τις διεθνείς συμβάσεις. Η διεθνής κοινότητα λοιπόν πρέπει να δράσει σωστά προς αυτή την κατεύθυνση και η Ιαπωνία θα συνεργαστεί μαζί της. Συνεπώς η Ιαπωνία θα επαναλάβει ξανά και ξανά τις αρχές της ελεύθερης ναυσιπλοείας και του κράτους δικαίου και θα επενδύσει και θα ερευνήσει στα πλαίσια οικονομικής συνεργασίας μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον για να πετύχουμε ευημερία και στήριξη στον τομέα της ασφάλειας, αλλά και συμμόρφωση προς το δίκαιο της θάλασσας με ό,τι μέτρα χρειάζονται και για την πρόληψη καταστροφών. Ενισχύοντας τη συνεργασία μας, η Ιαπωνία θα συντονιστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία, την Ινδία και την Ευρώπη. Και θα ολοκληρώσω το μήνυμά μου προς ε, τα μέλη της Κοβιτροπής σας ως εξής. Η Ασία και η Ευρώπη αντιμετωπίζουν κοινέ προκλήσεις σε σχέση με την ελεύθερη ε, διάβαση και την διεθνή τάξη. Πρέπει να δράσουμε σύμφωνα με τις κοινέ μας αξίες και αρχές, μεταξύ των οποίων ελευθερία, η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Οι προκλήσεις αυτές θα ισχύουν εφόσον οι Ηνωμένε Πολιτείε, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τρει δημοκρατικέ δυνάμει, θα συνεργαστούν μαζί. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ την εξοχότητά σα για τα όσα μα είπατε όσον αφορά του πυλώνε αυτού τη πολιτική ασφάλεια και άμυνα τη Ιαπωνία. Και τώρα, σίγουρα θα θέλετε να υπάρξει και ανταλλαγή απόψεων Οπότε, χωρίς άλλη καθυστέρηση, θα ζητήσω από τον Διευθυντή Βίγκαντ να πάρει το λόγο. Thank you very much. Uh, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την Επιτροπή που διοργάνωσε αυτή την ακρόαση. Χτες, με τα κράτη-μέλη έγινε ενδελεχής ε, συζήτηση περί της ασφαλείας στην Ασία. σύμφωνα με την στρατηγική, την παγκόσμια, δίνουμε, έχουμε δύο δράσεις στην ομολογήση. Πρώτα απ' όλα, να χαρτογραφήσουμε τη διασυνδημότητα και τα συναφή ζητήματα και ελπίζουμε αυτό να γίνει στρατηγική σχετική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά Θέλουμε μεγαλύτερη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την ειρήνη στην Ασία και να συνεργαζόμαστε και με του Ασιάτε εταίρου μα για θέματα ασφαλεία. Είναι βασικό στρατηγικό εταίρο μα η Ιαπωνία. Ο πρέσβή αναφέρθηκε επανειλημμένα στις στενέ σχέσεις που μας δένουν. Όλοι υπήρξαμε μάρτυρες των προσπαθειών από την Ιαπωνική πλευρά να ρυθμίσει το θέμα όταν επισκέφθη ο Πρωθυπουργό ο κ. Άμπε της Βρυξέλλες εν την προετοιμασία των συνόδων κορυφής G7 και G20. Επίσης θα ακολουθήσει και μια πολύ σημαντική διμερή σύνοδος κορυφής αργότερα αυτό το έτος. Είναι αναστατωμένο το διεθνές περιβάλλον και είναι πολύ σημαντική τώρα αυτή η συνεργασία. Περισσότερο ποτέ έχουμε κοινέ αξίες. Στηρίζουμε το κάτω δικαίου, την ελευθερία τη έκφρασης, τη φιλελεύθερη δημοκρατία και θέλουμε να έχουμε ένα λειτουργόν διμερές σύστημα βάσει προδιαγραφών και κανόνων. Η τελευταία σύνοδος κορυφής που έλαβε χώρα το 2015 καλωσόρισε την αυξανόμενη συνεργασία Ιαπωνία και Ευρωπαϊκή Ενώση στο τομέα της ασφαλείας και της ειρήνης. Συζητήσαμε και μελλοντική συμμετοχή της ε, Ιαπωνία σε ειρηνευτικέ αποστολέ. Μεταρρυθμίστηκε η πολιτική της Ιαπωνία στον τομέα αυτό και αυτό παρουσιάστηκε από τον κύριο Πρέσβη. Αν επιτρέπετε, θα εστιαστώ στον αντίκτυπο που θα έχει αυτή η μεταρρύθμιση σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια, όσον αφορά αυτό την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να υπάρξουν ειρηνικέ και σταθεροποιητικέ εξελίξει στην περιοχή. Δεν χρειάζεται να είναι κανεί ειδικό για την ασφάλεια στην Νοτιοανατολική Ασία για να δει ότι αυξάνονται οι εντάσει εκεί. Η Βόρεια Κορέα τακτικά κινείται με τρόπο που να απειλεί την Νότια Κορέα, την Ιαπωνία, την Κίνα και τη Ρωσία. και οι χώρες οι γειτονικές αναγκάζονται να καταφύγουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Οι εδαφικές διεκδικήσεις ίσως ε, να αναστατώσουν την περιοχή. Ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε, ο κ. Στήλισεν, είπε ότι όλα είναι πιθανά. Αυτό δείχνει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Όταν η Ιαπωνική κυβέρνηση ξεκίνησε ε, να ε, αλλάζει την πολιτική της για ασφάλεια, όλοι θεώρησαν ότι μπορεί να αυξηθούν οι εντάσεις. Πιστεύουμε όμως ότι αυτά που προτείνει η Ιαπωνική κυβέρνηση δεν θα αλλάξουν τη βασική θέση της Ιαπωνίας και του προσανατολισμού. Είπε ότι είναι φιλιρινική χώρα η Ιαπωνία, είπε ο κ. Πρέσβης. Τα τελευταία 70 χρόνια έτσι ήταν τα πράγματα. Και πιστεύουμε ότι έτσι θα συνεχίσει. Το νομικό πλαίσιο για στατιωτική παρέμβαση είναι άκρος περιοριστικό είναι πιο περιορισμένο από ό,τι για οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτό που ισχύει για την Ιαπωνία. Κυρίως όσον αφορά την χρήση δυνάμεων. Όπως και στη χώρα μου, απαιτείται κοινοβουλευτική σύμφωνη γνώμη. 1% του ΑΕΠ είναι θετικές δαπάνες. Αρκετά ενδιαφέρον να δει κανεί στον κόσμο τι γίνεται όσον φάτσα τι αμυντικέ διαπάνε. Αυτό είναι και κάτι που συζητάμε στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Το κοινό της Ιαπωνίας ε, δεν ε, διστάζει όσον αφορά την ανάπτυξη Ιαπωνικών δυνάμεων στο εξωτερικό και συζητείται το θέμα της παρέμβασης στο Νότιο Σουδάν. Ακούγονται πολλές επικρίσεις στην Ιαπωνία όσον αφορά αυτό το θέμα. Να Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τις παραμέτρους που επικρατούν στην Ιαπωνία, όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας. Πιστεύουμε ότι η χώρα θα παραμείνει πολύ συγκρατημένη και πολύ υπεύθυνη όσον αφορά τη χρήση ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχουν πολλές εδαφικές διεκδικήσεις και διαφορές. in Europe uh, already in the 70s and 80s. Um, and the most uh, obvious one is the one... Uh, λοιπόν, όπως γινόταν στην Ευρώπη στη δεκαετία του 70. Βλέπουμε και εδώ πόσο μας προσχολεί η Ρωσία και πόσο πολιτικό κεφάλαιο δαπανάται για την αντιμετώπιση του προβλήματος της Ρωσίας σε ύψιστο επίπεδο. Και εδώ υπάρχουν και διαφορές Ιαπωνίας-Ρωσίας όσον αφορά τις ε, βόρειες ε, περιοχές. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα ασφαλείας. Κυρίως αν λάβει υπόψη κανείς τις δυνατότητε που έχει η Βόρεια Κορέα όσον αφορά ε, βαλιστικούς πυράβλους με πυρηνικές κεφαλές. Το να, μπορεί να εκτοξεύσει πυρηνικές κεφαλές είναι πρώτη στην προτεραιότητα του καθεστώτος της Βόρειας Κορέας. Μας παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία που καταδεικνύουν την αύξηση του βεληνικού των πυράβλων της Βορείου Κορέας δεν είναι απειλή μόνο για τους άμεσους γείτονες της Βορείου Κορέας. Μπορούν να πλήξουν οι Βορειοκορεάτες και τις Ηνωμένε Πολιτείε. Και όχι στο απότερο μέλλον, αλλά πολύ σύντομα. Σε όλα αυτά η Κίνα αντιδρά και συνειδητά αποφάσισε να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες και να προωθήσει τα συμφέροντά της στην ε, νοτιοανατολική, στη θάλασσα της νοτιοανατολικής, στη νοτιοανατολική συνική θάλασσα μάλλον. Και αυτό ενισχύει την Ιαπωνία. Είναι αρκετά μετριοπαθής η ιαπωνική τοποθέτηση για την ώρα. αποφεύγει την κλιμάκωση των εντάσσεων στην περιοχή. Η αντίδραση των Ιαπώνων όσον αφορά τον επαναπροσωνατολισμό της αμυντικής τακτικής της χώρας ε, είναι μετριοπαθής. Δεν έγιναν αριζοσπαστικές ε, αλλαγές στην αμυντική τοποθέτηση της χώρας. Δεν έχει μόνο εταίρου στην Ανατολική Ασία αλλά και στην Νότια Ασία η Ιαπωνία. Υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός μεταξύ Ιαπωνίας και χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Αυτό οδηγεί σε πολυμερείς λύσεις για την ασφάλεια. Η θαλάσσια ασφάλεια δείχνει ότι έχουμε κοινά στοιχεία εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση με την Ιαπωνία μέχρι 50% του εξωτερικού εμπορίου περνάει από τον Ειδικό ωκεανό μέσω των στενών του Μαλάκα και πάει ε, στην θάλασσα της Νότιας Κίνας. Και αυτό μπορεί να έχει, ε, αν υπάρχουν προβλήματα, αρνητικές συνέπειες ε, για την οικονομία μας. Υπάρχει αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών και των εταιριών όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Πρέπει λοιπόν και να γίνουν προσπάθειες, να υπάρχει συνεργασία για να αντιμετωπιστούν οι παράγοντες ασταθείας. Καλωσορίζουμε συμμετοχή των ασιατικών εταίρων στην επιχείρηση Αταλάντα στο κέρας της Αφρικής μια κορεατική φρεγάτα συμμετέχει, άρχισε συμμετέχει σε επιχειρήσεις και ελπίζουμε σύντομα να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις ε, για ένα πλαίσιο συμμετοχής της Ιαπωνίας και να μπορούμε να συνεργαστούμε σε ε, αποστολές ασφαλείας μαζί με την Ιαπωνία όταν θα καθοριστούν οι όροι και θα υπάρξει συμφωνία. Έχουμε άλλες αιτικές χώρες που μας πλησίασαν πρόσφατα για την ασφάλεια στην ε, αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές. Η Ευρώπη ήταν πάντα παρούσα στον επιχειρηματικό τομέα. Έχει επίσης αναπτύξει θαλάσσιες ε, δυνάμεις, ε, ναυτικές δυνάμεις, αλλά δεν έχει την διαπαρουσία όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχουν 54.000 στρατιώτες Αμερικανοί στην Ιαπωνία. Και ε, υπάρχουν συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ για την ασφάλεια της Ιαπωνίας. Η νέα νομοθεσία περί ασφαλείας έχει πρόθεση να ενισχύσει τη συμμαχία ΙΠΑ Ιαπωνίας. Πρέπει να έχουμε επίγνωση αυτού. Δεν μπορεί να αντικαταστήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση της ΙΠΑ, αλλά υπάρχει ε, περιθώριο να αυξηθεί επιχειρησιακά η συνεργασία μας και με τους Ιάπωνες και με τους Ασιάτες εταίρους στην περιοχή. Έχουμε ε, κοινά συμφέροντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέλουμε να υποστηρίξουμε ειρηνευτικές διαδικασίες στην περιοχή, είτε αυτές είναι στις Φιλιππίνες, είτε στο Μιανμάρ, στη Σρι Λάνκα κατ' παρελθόν, στην Ινδονησία κατ' παρελθόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιείται σε του τομεί και έχουμε καλή συνεργασία με την Ιαπωνία όσον αφορά τα νέα προβλήματα ασφαλείας. Σε κάποιες χώρες ήταν γνωστά τα προβλήματα, θέλουμε να γίνουν περισσότερα και κλείνοντας λέγω ότι δεν θέλουμε να δείξει τη δύναμή της όσον αφορά την ασφάλεια στην Ασία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει συμβατική προσέγγιση για την ώρα στην Ασία. Πιστεύουν ότι ένα ισχυρό ναυτικό αρκεί. Ε, είναι και θέματα όμως άλλα. Κυβέρνο, ασφάλεια, ε, ριζοσπαστικοποίηση, ε, ακραίος, ακραία εξτρεμιστική τρομοκρατία. Χρειάζεται ευρύτερο ορισμός για την ασφάλεια. Προσπαθήσαμε να το κάνουμε αυτό παγκόσμια, στη στρατηγική μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι πολύ δραστήρια στους τομείς αυτούς η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεργασία με τον ΝΑΤΟ αλλά έχουν περισσότερες δυνατότητες στον τομέα αυτό από ό,τι έχει το ΝΑΤΟ. Παρέχουμε συνδρομή σε κατάλληλες δομές ασφαλείας που ίσως να προσελκύουν ασιάτες εταίρους μας, κυρίως το ΑΖΕΑΝ, αλλά δεν είναι κάτι που αφορά απλώς στατητικές δυνάμεις, οι οποίες βέβαια παίζουν σημαντικό ρόλο. Η δεύτερη καινοτομία τρόπο αντιμετώπιση Ευρώπης και Ασίας είναι πώς μπορούν να συμβάλλουν περισσότερες ηθικέ χώρες όσον αφορά τα αμυντικά συμφέροντα της ε, ε, Ευρώπης που ίσως να συμφέρουν αυτές οι προσεγγίσει και την Ασία. Χρειάζεται αμοιβαία ε, προσέγγιση. Έχουμε οικονομική αλληλεξάρτηση και η ασφάλεια της Ασίας ίσως να εξαρτάται και από την οικονομική ευημερία της Ευρώπης και αντιστρόφως. Άρα θα θέλαμε να δούμε πιο συγκεκριμένες προσπάθειες που θα καταβάλλονται με τη συνεργασία των ασιατών εταίρων. Ίσως έχουμε προχωρήσει περισσότερο με την Ιαπωνία όσον αφορά την άμεση συνεργασία, είτε είναι στη Μέση Ανατολή, είτε είναι στην Αφρική. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Ευχαριστώ πολύ το Διευθυντή Βίγκαντ και τώρα η κυρία Τερίζα Φαλών. Έχετε το λόγο κυρία μου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ. Συγγνώμη για τη φωνή μου, είμαι πολύ κρυωμένη. Ήμουν στο Eurostar, καθόμουν δίπλα σε κάποιον που έβηχε συνέχεια χωρίς προφύλαξη και με κόλλησε. Λοιπόν, ε, θέλω συγχαρώ τους δύο προηγούμενους ε, ομιλητές ε, και τον ε, πρεσβευτή Κοντάμα για την εξαιρετική παρουσίαση και για τα σχόλιά του συγχαίρω τον κύριο Βίγκαντ. Λοιπόν, θα δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα μέσα από ένα άλλο πρίσμα. πρόσφατες τάσεις της σινοϊαπωνικές σχέσεις σε σχέση με την Ανατολική Συνική Θάλασσα, σε ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο, υπάρχει πρόοδος προς ένα μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων. Εδώ έχουμε τις περιοχές ε, που απασχολούν την Ιαπωνία, ε, στην ε, Νότια και την Ανατολική Κινέζικη θάλασσα και στη Βόρεια Κορέα υπάρχουν προβλήματα, είναι δύσκολη περιοχή Τώρα, για το ιστορικό, το εθνικό αφήγημα ταπείνωσης, 100 ε, χρόνια διέρχεση η Ιαπωνική ταπείνωση, είναι σημαντικό αυτό για την εξωτερική πολιτική, γιατί ε, ε, επηρεάζονται πολλές δραστηριότητες σήμερα στην περιοχή από το παρελθόν. Λοιπόν, η φιλιρινική διπλωματία του Πρωθυπουργού Άμπε, η Κίνα γίνεται πιο επιθετική, η, στρατιωτικοποιείται η Βόρεια Κορέα, ε, υπάρχει πρόβλημα τώρα με τον Τραμπ και την, την απέτησή του για ε, επιμερισμό των βαρών. ε, υπάρχει η αναθεώρηση του συντάγματος, η νέα ερμηνεία του συντάγματος πιο ε, εκτατική. Το 2012 χαράκτηκε η Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια και ε, βάθινε η συνεργασία σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ Ιαπωνίας και Ηνωμένων Πολιτειών ε, και οι εξαγωγές όπλων συμπεριέλαβαν και το ΑΣΕΑΝ. Υπάρχει λοιπόν αύξηση των στρατιωτικών ε, δραστηριοτήτων γύρω από πολλά νησιά στην περιοχή. Είδαμε και τις διαφάνειες του πρέσβη σχετικά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ατυχήματα, κακούς υπολογισμούς. Τώρα, τι έγινε το 2015. Αυτή ήταν μια ε, κίνηση αντι-Ιαπωνική σε σχέση με τα 70 χρόνια την επέτειο από το τέλος του πολέμου. Ε, εδώ ε, γίνονται προσπάθειες από την Κίνα να επηρεαστεί ο λαός αρνητικά απέναντι στην ε, Ιαπωνία. Είχαν σημειωθεί πολλές δραστηριότητες το 2013 να σας θυμίσω ότι η Κίνα στην Ανατολική Κινέζικη θάλασσα ε, δήλωσε ότι υπάρχει ε, αμυντική ζώνη ε, ντοπισμού. το 2000, από το 2012 άρχισαν αυτά. Επίσης ε, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις όπου εισήλθαν στα ιαπωνικά χωρικά είδα τα κινέζικα σκάφη, παραβιάσεις ε, ε, θα, και ε, θαλάσσιες και εναέριες. Ο αμυντικός προϋπολογισμός σε, από τεχνικής άποψης μειώνεται, ε, αλλά εδώ βλέπετε το 2000 σε σχέση με το 2015 συγκριτικά την κατάσταση. Τώρα έχουμε ε, περισσότερες δαπάνες στον τομέα των εξοπλισμών και κυρίως στην αυπήγηση νέων πλοίων. Καινούριε φρεγάτες, καινούργια αντιτορπιλικά, σύγχρονα. Ε, εδώ με γεωμετρική πρόοδο αυξάνονται οι δαπάνες. Ε, εδώ ένα σκάφος της ακτοφυλακής 10.000 τόνων, τεράστιο. Είναι για την ακτοφυλακή, δηλαδή ε, ε, κάνει περιπολίες εκεί, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αλλού. Ε, εδώ έχουμε τα πλοία της Κίνας που είναι η ακτοφυλακή, τα σκάφη που χρησιμοποιούνται στον ε, πόλεμο. Η ακτοφυλακή μειώνει το στρατιωτικό τους αποτύπωμα γιατί καλύπτει ε, δυνητικά στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μιλάμε για μια γκρίζα ζώνη εδώ. Ε, είναι κάτι παρόμοιο με τις επιχειρήσεις που έχουμε δει και αλλού στην Κρυμαία κλπ. Η διεθνής κοινότητα αντέδρασε στην Κρυμαία. Η Κίνα παρακολουθεί προσεκτικά να δει πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και πώς θα αντιδράσει η Δύση, η ε, για να προσαρμόσουν ανάλογα τις δικές τους ε, κινήσεις. Ο πρεσβευτής μίλησε για τη Βόρεια Κορέα, το ΘΑΝΤ, ε, αυτή το χερσαίο σύστημα βαλιστικής άμυνας των Αμερικανών. Ε, αυτή είναι μια προοπτική που μπορεί να δημιουργήσει σφοδρές αντιδράσεις, δηλαδή ούτε η ε, Κορέα ούτε η Κίνα βλέπουν με καλό μάτι αυτές τις εξελίξεις. Εδώ βλέπ, γνωρίζετε τις εντάσεις στην περιοχή της Νότιας Συνικής θάλασσας. Τον Ιούλιο το Παγκόσμιο Διαιτητικό Δικαστήριο έλαβε μια απόφαση ε, περιορίζοντας την ε, Κίνα. Ε, εδώ βλέπετε τις βραχονισίδες Σκάρμπορο. Είχαμε το 2012 προβλήματα με την ακτοφυλακή των, της Ινδονησίας. Ε, εδώ ε, είχαν γίνει επιχειρήσεις που κατέστρεψαν ε, το περιβάλλον διότι χτύπησαν το, το, και κατέστρεψαν τους, τους υφάλους στην περιοχή. Οι Κινέζοι έμειναν εκεί παρόλο που υπήρξαν σήματα για αποχώρηση των δυνάμεων από την περιοχή λόγω επερχόμενου τυφώνα. Εφτά οι ύφαλοι ή τεχνικές νησίδες όπως και αν ε, περιγραφούν, σχηματίζουν 7 νησίδες στην περιοχή. Το Βιετνάμ, η Μαλαισία ε, κάνουν παρόμοιες κινήσεις, αλλά κανένα κράτος δεν προχώρησε στην κλίμακα ε, στην οποία προέβη η Κίνα πριν παρέμβει το Διαιτητικό Δικαστήριο. Και βλέπετε εδώ τη μεγάλη αλλαγή, τη στρατιωτικοποίηση επίσης των νησίδων αυτών πράγμα που αλλάζει τελείως το φυσικό χώρο στην περιοχή. Τώρα, γιατί παλιά θεωρούσαν ότι αυτές οι νησίδες μπορεί να καταστραφούν πολύ γρήγορα. Τώρα όμως έχουν αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Φαίνεται αυτό και στην διαφάνεια. Έχει αλλάξει η άρδινη εικόνα της περιοχής. Η, στην νότια Κινέζικη θάλασσα. Γιατί είναι τόσο σημαντική. Οι τελευταίες ε, ψηφίδες είναι οι βραχονισίδες Κάρμπορο. Η Κίνα είπε ότι θα δημιουργήσει ένα κέντρο ε, δοκιμών περιβαλλοντικών εκεί. Αυτό το έχει κάνει προηγουμένως και σε άλλες νησίδες και θα το επαναλάβει. Και είναι η τελευταία ψηφίδα. Εάν έχουν έλεγχο αυτής της περιοχής θα ελέγχουν ολόκληρη την περιοχή. Ε, και θα μπορεί να λειτουργήσει αυτή η αερία ε, ε, αμυντική ζώνη που θέλουν να δημιουργήσουν για τον εντοπισμό ξένων σκαφών. Ο Πρωθυπουργό Άμπε είναι ακούραστο στις προσπάθειες που κάνει για την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Προσπαθεί να αποκαταστήσει επίσης διπλωματικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες. Όλα αυτά τι σημαίνουν για την Ευρώπη, γιατί μας ενδιαφέρει εμάς, τι γίνεται με τους Ευρωπαίους μετά την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Ε, είμαι περήφανη διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε χωριστή δική του δήλωση Βλέπουμε αύξηση των κινέζικων επενδύσεων στην Ευρώπη. Πώς ορίζουμε την οικονομική δύναμη της Κίνας, ε, ε, αντιμετωπίζεται με ε, διάφορους τρόπους σε οικονομικό επίπεδο, με εμπορικές κυρώσεις. Βλέπουμε επίσης βλέπουμε τις τεράστιες επενδύσεις στην Ευρώπη, ενώ το αντίστροφο είναι δύσκολο, δηλαδή ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Κίνα. Η Τράπεζα Επενδύσεων που έχει δημιουργηθεί. Τώρα όλη αυτή η οικονομική επιρροή πώς ε, μεταφράζεται συγκεκριμένα. Ε, στη Κροατία είχε μια διαφορά με τη Σλοβενία. Η, η Ελλάδα έχει δεχθεί στο Μπειραιά πολλές επενδύσεις. Η Ουγγαρία επίσης είναι μελλοντικός επενδυτικός στόχος. Ε, αντί να ε, χαιρετήσει την απο... ή να στηρίξει την ε, δήλωση του Διαιτητικού Δικαστηρίου οι Ευρωπαίοι απλώς την έλαβαν υπόψη, δηλαδή δήλωσαν ότι έλαβαν γνώση. Ε, δεν δήλωσαν τις, ότι συμφωνούν. Ε, βλέπετε εδώ τη στρατηγική της Κίνας από τον, από τον Πειραιά μέχρι τη Βόρεια Ευρώπη. Η Ευρώπη είχε μια μεγάλη ευκαιρία να στηριχθεί στο διεθνές δίκαιο και να το στηρίξει με την, από την, επίσης αποστέλλοντας έτσι ένα ηχηρό μήνυμα στην Κίνα και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Κίνα έχει ένα χρονικό ορίζοντα τη, τη, τη, θέλουν ε, να ε, ανασυγκροτηθούν, θέλουν να αποκτήσουν ε, την Ταϊβάν πίσω. Ε, ε, καλό είναι να μιλήσουμε όμως εδώ για την Ιαπωνία, γιατί η ακρόαση για την Νότια και την Ανατολική Συνική Θάλασσα θα γίνουν μετά. Οπότε εδώ θα πρέπει να δώσετε τα συμπεράσματά σας, να προλάβουμε να κάνουμε και συζήτηση και να ακούσουμε τις ερωτήσεις. Λοιπόν, για να κλείσω ανεξάρτητα από τη θέση της Ιαπωνίας αντιδρούν στα τεκτενόμενα στην περιοχή. Η κινέζικη οικονομία επιβραδύνεται και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την κρίση στην Ανατολική Συνική Θάλασσα. Ακόμα και αν έχουμε έλεγχο και διαχείριση της κρίσης, είναι δύσκολο να ε, έχουμε αποκλιμάκωση. Ε, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα έστω και αθέλητα. Ε, επίσης, ε, η εθνική στρατηγική της ε, Κίνας ε, ε, μπορεί, αν ολοκληρωθεί, να δημιουργήσει πιο συγκροτημένη πολιτική. Ή ο κίνδυνος ατυχήματος μπορεί να είναι υψηλότερος από ό,τι θεωρούν πολλοί. Επηρεάζεται η Ευρώπη από τις εξελίξεις εκεί. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και περιμένω τις ερωτήσεις σας. Okay, madam. Once more, I'm very sorry. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη που σας διέκοψα πριν, αλλά αυτό το θέμα είναι το θέμα της ακροασής μας. Ε, γι' αυτό ήθελα να επικεντρωθούμε τώρα στην Ιαπωνία. Τέιπ ό,τι έχει να κάνει με την Ιαπωνία λοιπόν συζητάμε τώρα παρόλο που τα θέματα αυτά σίγουρα ε, παίζουν ρόλο και στο επόμενο θέμα μας. Αλλά τώρα μας ενδιαφέρει η μας ενδιαφέρει μεταρρυθμίσεις της Ιαπωνίας. Λοιπόν, ο λόγος του συναδέρφους. Παρακαλώ ότι σχόλια έχετε παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά που ακούσατε τον κύριο Κοντάμα, τον κύριο Βίγκαντ και την κυρία Φαλόν. Ο κύριος Πασκού θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Γνωρίζω ότι η υποεπιτροπή μας ετοιμάζει την επίσκεψή της στην περιοχή. Το ξέρετε. Αλλά ελπίζω η συζήτηση αυτή που κάνουμε να μην γίνεται μόνο γι' αυτό. Χαίρομαι λοιπόν για την πρωτοβουλία που πήρατε να συζητηθεί αυτό το θέμα γιατί είναι ένας ε, τομέας που μπορεί να επηρεάσει την ειρήνη και την ασφάλεια ολόκληρου του συστήματος. Γι' αυτό και οι σχέσεις στην περιοχή Μα ενδιαφέρουν όλου ιδιαίτερω. Και χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία λοιπόν σήμερα να συζητήσουμε την προσέγγιση της Ιαπωνία όσον αφορά την ασφάλεια και την αμυνά τη και να τη συζητήσουμε με τους Ιάπωνες φίλους. Αναφερθήκατε στην αποτροπή που είναι η Αμερικανική-Ιαπωνική Συμμαχία. όντω ε, είναι μια δύναμη αποτροπής, συγχρόνως όμως απαιτεί και έναν ε, λογικό εταίρο. Έτσι. Χρειάζεστε λογική και από την άλλη πλευρά. Και φοβάμαι, βλέπετε, ότι δεν υπάρχει αυτό από την πλευρά της Βόρειας Κορέας, αυτή η λογική. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην άμυνα, γιατί όταν η αποτροπή δεν λειτουργεί, δεν ε, φέρνει αποτελέσματα, πρέπει να περάσουμε στην άμυνα. Θα ήθελα λοιπόν να γνωρίζω, διαβάσαμε τα μέτρα που παίρνετε, ωραία, αλλά θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η εκτίμησή σας Τι άλλο θα χρειαστεί ναι. αν η αποτροπή δεν φτάνει ή τι άλλο χρειάζεται. Και τι γίνεται όσον αφορά την οικονομική εκμετάλλευση του βόρειου τμήματος. Πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο παγίωσης δηλαδή σε αυτήν την τόσο περίπλοκη κατάσταση. Να υπάρχει ένα σταθεροποιητικό παράγοντα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Πασκού. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο εδώ, γιατί δεν έχω εγώ κανέναν άλλο στον κατάλογό μου. Κάποιος άλλο θέλει να μιλήσει. Ο κύριος Μπέλετ. Όχι, εντάξει, ο κύριος Μπουστινάρο, ούτε. Καλώς. Όλες αυτές τις αγωγικές ε, παρατηρήσεις που ακούσαμε, οι παρουσιάσεις ήταν ξεκάθαρες, συνεπώς. Λοιπόν, όλοι μας γνωρίζουμε αυτόν τον ανατολικό παράγοντα και τη σημασία που έχει για την παγκόσμια ασφάλεια. Και κυρία Φαλό, πολύ εκτιμήσαμε και τις δικές σας παρατηρήσεις σχετικά με πολιτικές που ακολουθεί η Κίνα και ότι πρέπει να τις έχουμε και αυτές οι υπόψεις μας για να έχουμε ολόκληρη την εικόνα. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον πρέσβη κάτι για την δικιά του εκτίμηση όσον αφορά την ανάπτυξη ε, πολιτικών στις Φιλιππίνες. Ποιες είναι οι προοπτικές για τις σχέσεις Ιαπωνίας με τις Φιλιππίνες. Ποιες είναι οι δυσκολίες, ποιες είναι οι προκλήσεις και ποιες είναι οι προσδοκίες που έχετε. Ξέρω ότι υπήρξαν κάποιες προτάσεις για επισκέψεις. Μας, μας απασχολούν οι εξελίξεις στις Φιλιππίνες για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η χώρα αυτή είναι σημαντική για την ασφάλεια και γενικά τις εξελίξεις στην περιοχή. Γι' αυτό δεν θα σας ρωτήσω τίποτα άλλο, ίσως ένα δεύτερο γύρο. Αλλά θέλω να αφήσω περιθώρια και για να κάνω ερωτήσεις και στο επόμενο πάνελ που θα έχουμε για την ακροασή μας δηλαδή. Ο πρέσβης, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα απαντήσω στις δύο ερωτήσεις του κύριου Πασκού και πρώτα απ' όλα για τις προσπάθειες της Ιαπωνίας, τις αμυντικές, για να ανταποκριθεί σε στρατιωτικές απειλές και τη... τις πυρηνικές δυνατότητες που έχει η Βόρεια Κορέα. Λοιπόν, η Ιαπωνία διατηρεί τη συμμαχία με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Δηλαδή, μέχρι τώρα πιστεύουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες εξακολουθούν να παίζουν ένα ρόλο ασπίδας για μας. Πρέπει να συνεχίσουμε λοιπόν να βασιζόμαστε στις δυνατότητες προστασίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν ο Πρωθυπουργό Άμπε συναντήθηκε με τον κύριο Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο Πρωθυπουργό έπεισε τον κύριο Τραμπ για την μεγάλη σημασία που έχει αυτή η συμμαχία Ιαπωνία Ηνωμένων Πολιτειών για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Και ο κύριος Τραμπ μας διαβεβαίωσε ότι συμφωνεί κάτι το οποίο ήταν ανακούφιση για μας. Τώρα όσον αφορά την ε, Βόρεια Κορέα, υπάρχει μια ηρωνία. Ο, ήταν ε, ακριβώς στο Μαλάκο στην ε, Φλόριντα ο κύριος Τραμπ με τον πρωθυπουργό μας τον κύριο Άμπε και τότε ακριβώς ήταν που έπεσε ο δεύτερος ή ο τρίτος βαλιστικός πύραυλος. Και ήταν μια καλή ευκαιρία για να συνειδητοποιήσει ο κύριος Τραμπ τι συμβαίνει. Συνεχίζουμε να βασιζόμαστε στις αμερικανικές δυνάμεις, αλλά συγχρόνως αναπτύσσουμε και εμείς και ενισχύουμε τα δικά μας αμυντικά συστήματα με τη βοήθεια των ΗΠΑ. Για τη Ρωσία. Θέλω να πω ότι με τη Ρωσία η συμμαχία παραμένει, όπως είπε και ο κύριος Βίγκαν, υπάρχει σταθερότητα όλα αυτά τα χρόνια. Ο κύριος Άμπε ανέλαβε πρωτοβουλία να έρθει σε επαφή με τον κύριο Πούτιν και του είπε να προσπαθήσουμε να έχουμε μια νέα προσέγγιση που να βασίζεται στην πεποίθηση, που είναι πεποίθηση του Πρωθυπουργού και που δεν είναι βέβαια κάτι εύκολο, αλλά και θα σας το πω με τη δικιά μου διατύπωση, να δημιουργήσουμε κάποια αποτροπή να δούμε ποιες είναι οι εδαφικές διενέξεις και να βρούμε μια νέα προσέγγιση που να βασίζεται σε κοινέ οικονομικές δραστηριότητες από τις οποίες να μπορούν να αποφεληθούν και οι Ιάπωνες και οι Ρώσοι στα διαφελονικούμενα νησιά. Φυσικά πρέπει να λυθεί το θέμα του ποιονού δικαιοδοσία είναι. Ποιος νόμος εφαρμόζεται, ο Ιαπωνικός, ο Ρωσικός. Καταλαβαίνω ότι αυτό μπορεί να είναι εμπόδιο. Γι' αυτό όμως πρέπει να βάλουμε τη φαντασία μας να δουλέψει. Και αυτό κάνουμε. Τώρα για να απαντήσω και στην ερώτηση της Προέδρου για την Ιαπωνία και τις Φιλιππίνες. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τις Φιλιππίνες καλύτερες από ποτέ. Και εξαιτία της μακράς ιστορία των Φιλιππίνων που έχουν μια πολύ γερή και καλά λειτουργούσα δημοκρατία με τα πάνω και τα κάτω, αλλά πάντως και η οικονομία τους επίσης είναι εύρωστη. Ξέρετε ότι πήγανε οι Φιλιππίνες στο δικαστήριο και στη Χάγη ε, συζητήθηκε ε, το θέμα για τις εκδικήσεις της Κίνας και ξέρετε ότι το δικαστήριο δικαίωσε τις Φιλιππίνες. Έτσι λοιπόν και εμείς στηρίξαμε την απόφαση αυτή και ενθαρρύνουμε τις Φιλιππίνες να βασιστούν στην προσέγγιση αυτή από κοινού με τους εταίρους από τις χώρες ΑΣΕΑΝ. Η ΑΣΕΑΝ με την Κίνα πρέπει να καταλήξουν σε έναν κώδικα δοντολογίας. Νομίζω πάντως ότι μεταξύ των χωρών ΑΣΕΑΝ φυσικά υπάρχει κάποια διαβάθμιση όσον αφορά τις σχέσεις τους με την Κίνα και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμβαίνει αυτό. Αλλά βασικά είμαι αισιόδοξο και να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τις Φιλιππίνες. ευχαριστώ. Πρόεδρος, σε ευχαριστούμε πολύ εξοχότης. Τώρα σας παρακαλώ εσάς, κυρία Βίγκαντ. Well, I would like to um, emphasize that uh, in... Uh, Θέλω να τονίσω ότι όσον αφορά την Ασία και τα θέματα ασφαλείας η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ρόλο. Είναι προφανές για αυτούς που δουλεύουν σε ομάδες προβληματισμούς αλλά όχι και για τις ομάδες προβληματισμού και τους δημοσιογράφους στην Ασία. Θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ουσιαστικά ε, μια συνάθρηση ε, ισχυρών κρατών. Υπάρχουν ιστορικοί και πολιτισμικοί δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικό προνόμιο στην περιοχή μας είναι η ισχύς του ιδιωτικού τομέα σε όλη την περιοχή. Η Ευρώπη είναι υπαριθμόν ένας εταίρος ή εταίρος υπαριθμόν δύο για άλλες χώρες είτε όσον αφορά το εμπόριο ή επενδύσεις. Και η αύξηση, η ανάπτυξη μάλλον της Κίνας που ξέφυγε από την φτώχεια δεν θα συνέβαινε χωρίς τις μαζικές επενδύσεις των ευρωπαϊκών εταιριών στην Κίνα. Χωρίς την πρόσβαση στην αγορά που είχε η Κίνα. Μετά τις σημαντικές εξελίξεις στην Ιαπωνία με το Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο που ήταν παράλληλη, μια παράλληλη εξέλιξη με την άνοδο της ε, Ευρώπης που ξαναγεννήθηκε τις τάχτες της. Παρόμοια πράγματα συμβαίνουν σε πολλές χώρες του ΑΖΕΑΝ που έχουν πολύ ψηλό ρυθμό ανάπτυξης. Το ίδιο και ε, με την Ινδία. Αυτά δείχνουν ότι η Ευρώπη θεωρείται από εκεί σαν πάροχος ευημερίας ανάπτυξης, εμπορίου, επενδύσεων. Όπως ξέρετε, εσείς που εργάζεστε εδώ, η Ευρώπη είναι κάτι παραπάνω από αυτά και ανησυχίες για την εσωτερική ασφάλεια και την εξωτερική ασφάλεια έχουν προβληθεί για τους πολίτες. Όχι μόνο οι ανησυχίες, αλλά έχουμε και αιτήσει για αποτελεσματικότερη Ευρώπη. Και αυτά που συμβαίνουν στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια και στη Βόρεια Αφρική, στην Ανατολική Ευρώπη, επηρεάζουν την ασφάλεια της Ευρώπης και τα συμφέροντα επίσης και των εταίρων μας της Ασίας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια στοιχεία σταθείας στην Ασία επηρεάζουν τα οικονομικά μας συμφέροντα εκεί. Γι' αυτό θα πρέπει να συμμετάσχουμε, να ενεργοποιηθούμε περισσότερο, να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας και βεβαίως οι πιο προφανείς εταίροι μας για την εξωτερική πολιτική και διαμόρφωση πολιτική στην περιοχή είναι εκείνοι που συμμερίζονται τι αξίε μα, που έχουν παρόμοια νοοτροπία. Και η Ιαπωνία είναι στην πρώτη ε, θέση. Η Προέδρος στην αρχή έθεσε ένα ερώτημα για το θέμα της παγκόσμιας κατάστασης. Χρειάζεται μια πλήρης προσέγγιση ολιστική, όχι μόνο απομονωμένα εμπορική πολιτική, απομονωμένα επιταξιδική πολιτική, η ασφάλεια, η ανάπτυξη, η εξωτερική πολιτική, όλα μαζί, σφαιρικά, αποτελούν ένα σύνολο και κάνουν τη διαφορά. Γι' αυτό ε, επεκτείνουμε, λοιπόν, τη συνεργασία μας θέματα ασφαλείας με τους εταίρους στην Ασία. Έχουμε πολλές χώρες στην περιοχή και η Ιαπωνία πρωτίστως έχει ευρύτερα συμφέροντα και πέρα από αυτή την κοντινή περιοχή θέλουμε να συνεργαστούμε μαζί με την Ιαπωνία. Για τη διαχείριση των κρίσεων, πρόληψη συγκρούσεων, υποστήριξη ειρηνευτικών διαδικασιών, καταπολέμηση νέων απειλών για την ασφαλειά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυντά, κύριε Βίγκαντ. Πριν δώσω το λόγο στην κυρία Φαλών, θα ήθελα να ερωτήσω και κάτι. Αν ο κύριος πρέσβης έχει την καλοσύνη να προσθέσει κάτι με τα χαρά θα ήθελα να τον ακούσω. Κυρία μου, αναφερθήκατε στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων. Σε προηγούμενες συζητήσεις στην Επιτροπή, σήμερα, νωρίτερα, κουβεντιάσαμε την πολιτική άμυνας και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Και εγώ έθεσα το ζήτημα του ρόλου του δολαρίου σαν νόμισμα για αποθεματικό σε παγκόσμια κλίμακα. Πώς αξιολογείτε αυτή την πρωτοβουλία στα πλαίσια της παγκόσμιας νομισματικής τάξης. Κάτι που σχετίζεται άμεσα και με θέματα σκληρής ούτως υπήν ασφαλείας. Υπάρχουν κάποιες πτυχές προς εξέταση. Και ίσως κύριε Πρέσβη, αν θα μπορούσατε να αναφερθείτε κάπως σε αυτό και στην κατάσταση Γενικά στην κατάσταση που στον κόσμο θα μας βοηθούσε. Κυρία μου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να επανέλθω γρήγορα στην αρχική σας ερώτηση για τις Φιλιππίνες. Ένα κλασικό δίλημα είναι αυτό. Λοιπόν, κέρδισαν στο δικαστήριο. Τα πήρε όλα. Τα πήραν όλοι στην εκδίκαση των διενέξεων των Φιλιππινών με τις, ε, των Φιλιππίνων με την Κίνα. Αυτό είναι το δίλημα που έχουν οι μεγάλες χώρες και οι μικρές χώρες. Οι Φιλιππίνες νίκησαν μεν στο δικαστήριο, όμως τελικά αποφάσισαν όσον αφορά τα εδαφικά να προσπαθήσουν να συνοηθούν με την Κίνα λοιπόν σταδιακά προχωρούν προς τις υφάλου. σταδιακά κάνουν σαλαμοποίηση όσον αφορά την προσέγγιση οι Κινέζοι και προχωράνε στι διεκδικήσει του. Και είναι δύσκολο να απαντήσει αυτό. Είπαν οι Φιλιππινέζοι λοιπόν ότι δεν μπορούν να προστατεύσουν αυτή την περιοχή. Έχασαν. Έχασαν ολόκληρη περιοχή. Δεν ξέρω αν αυτό δείχνει τι θα γίνει και στι υπόλοιπε περιοχέ τη χώρα και τα άλλα κράτα που δεν μπορούμε, είναι πολύ μεγάλη δύναμη η Κίνα και τελικά όλοι θα πρέπει να λυγίσουμε. Όσον αφορά σχέσεις Ιαπωνίας-Φιλιππίνων, ήταν πάντα δραστήρια η Ιαπωνία ε, όσον αφορά την ανάπτυξη ε, συνεργασίας με τις Φιλιππίνες, όσον αφορά και την έλεγχο των θαλασσών κλπ. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να το υποστηρίζει. Με την νέα κυβέρνηση Τραμπ επικρατεί το χάος. Πρέπει να παρέμβει και να καλύπτει το κενό Ευρωπαϊκή Ένωση και να υποστηρίξει την τήρηση των διεθνών προδιαγραφών. Αυτή την ε, περίοδο αβεβαιότητας και χάους που άρχισε να επικρατεί με την κυβέρνηση Τραμπ. Έχετε δουλειά να κάνετε και ελπίζω να τα καταφέρετε. Τώρα, όσον αφορά τις επενδύσεις, έχουμε την πρωτοβουλία ε, για το μονοπάτι του μεταξύ, όπως αποκαλείται. Ε, είναι το θέμα της διασυνδυσιμότητας να ενωθούν οι καρδιέ, οι λαοί κλπ. Αυτή είναι η πρωτοβουλία, αυτό αφορά η πρωτοβουλία. Και, θέλουμε και θέλουν το Ιωάννα να γίνει διεθνέ νόμισμα. Και το δούνου του το έβαλε στο καλάθι του εμπορίου, αλλά όταν υπάρχει κρίση δεν προσφεύγει ο κόσμο στο Ιωάν, αλλά στο δολάριο. Θα είναι πολύ δύσκολο να αντικατασταθεί, ίσω να συμβεί τελικά, αλλά αυτή είναι η μεγάλη στρατηγική τη κίνα και ελπίζουν να το καταφέρουν. Έκανα έρευνα λοιπόν για το θέμα αυτό δεν είπαν ότι πιστεύουν σε αυτά τα κάτι μελη Στον Ηνωμένο Βασίλειο ε, δώσανε δικαιώματα εμπορικά στο Ιουάν. Πήραν το μήνυμα σε διάφορες ε, χώρες. Έχουν αυτή τη στρατηγική. Ξέρουν από ιστορία. Προσπαθούν λοιπόν να κινηθούν σωστά για να επεκτείνουν την ισχύ τους οι Κινέζοι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι κύριε Πρέσβη και μετά θα δώσουμε το λόγο στον κύριο Μποστινάρου, θα είμαι πολύ σύντομο για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων. Λοιπόν, ε, οι ΙΠΑ θεωρούνται τελικά ότι είναι το μαύρο πρόβατο, ότι έχουν φύγει από το κοπάδι. Εμεί δεν μπήκαμε στην Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων. Κοιτάξτε, ποια είναι η πραγματικότητα κατά την άποψή μου. Η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων υποτίθεται ότι θα παρέχει διεθνή δανειοδότηση για εμπορικού σκοπούς. Πόσοι από εσά γνωρίζετε πλήρως τι ακριβώς συμβαίνει, Πώς, πόσα προγράμματα που χρηματοδοτηθούν από τράπεζα έχουν εντοπιστεί και έχουν εγκριθεί από την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και έχουν υλοποιηθεί. Εγώ δεν βλέπω να υπάρχουν πολλά. Πιστεύω λοιπόν ότι άλλο η ιδέα και άλλο η πράξη. Είναι εντελώς διαφορετικό αυτό. Το γνωρίζουμε. Από ε, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ασιατική Τράπεζα, την Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων πολλές εμπειρίες. Εγώ έχω εμπλακεί στα προγράμματα ε, ενισχύσεων κλπ. Τι θέλω να πω. Λοιπόν, είναι Θέλει μεγάλη προσπάθεια η χορήγηση βοήθειας. Δεν θέλω να είμαι Δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Και αυτό αντιμετωπίζει τώρα η Σετική Τράπεζα Επενδύσεων. Λοιπόν, για το θέμα αυτό της Κίνας, να πω κάτι. Πέρσι, η Κίνα με το Σιν Πιν έχει θεσπίσει τους ε, ελέγχους των ε, κεφαλαίων, capital controls. Προσπαθεί να αποφύγει τη διαρροή κεφαλαίων από την Κίνα να μην πάνε τα κεφάλαια στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό αντιβαίνει της θέσεως που θα μπορούσε να δοθεί σε κάποιον αν θέλει τελικά το νόμισμά του ε, να γίνει διεθνές νόμισμα. Η Κίνα αυτοπυροβολείται που θέλει να γίνει, να έχει ένα διεθνές σεβαστό νόμισμα. Το Ιωάννα γίνει διεθνές νόμισμα, θα δούμε συνεχίζει να αναπτύσσεται η Κίνα. Ο όγκος εμπορικών συναλλαγών θα εξακολουθεί να αυξάνεται. Και ούτω τρόπος ίσως τελικά να επικρατήσει και το, να διευρυνθεί ο ρόλος του κινέζικου νομίσματος όσον αφορά τις συναλλαγές. Ευχαριστώ εξοχότατε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Μπουστινάρου, θα ήθελα να κάνω Μία παρατήρηση σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Φαλόν για την ε, ασφάλεια στην Ανατολική Ισηνική θάλασσα. Ένας ομιλητής ε, θα κάνει μια σύντομη ομιλία σχετικά με διεθνή νομικά θέματα γιατί ειδικεύεται στο, δίκαιο, στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Οπότε θα ξαναγυρίσουμε στο θέμα αυτό. Δεν είναι αυτές οι συναντήσεις χωριστές πρωτοβουλίες. Η περιοχή αυτή μας ενδιαφέρει. Θα υπάρξει και αποστολή στην Ιαπωνία άλλωστε. Και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε συνέχεια στα θέματα αυτά. Ο κ. Μπουστινάρου, ευχαριστώ. Είναι βέβαιο ότι η περιοχή του Ειρηνικού γίνεται η μεγαλύτερη οικονομική περιοχή παγκοσμίω. Είναι μεγάλη αλλαγή. Τη βλέπουμε όλοι όμως. Βέβαια, το αβέβαιο εκτός από τις άλλες αβεβαιότητες τακτικής και στρατηγικής είναι ότι με την απόφαση του Τραμπ να αποσύρει την υπογραφή του από τη συμφωνία TPP η περιοχή αυτή, αν θέλετε, υπέγραψε το πιστοποιητικό θανάτου του TPP. Τι πιστεύετε, πώς θα εξελιχθούν οι εμπορικές σχέσεις στην περιοχή του Ειρηνικού σήμερα και ποιος θα υποκαταστήσει το κενό που αφήνουν. Μπορεί δηλαδή ο ειρηνικός να γίνει εμπορική περιοχή υπό την ηγεμονία της Κίνας γιατί όλα αυτά δεν έχουν να κάνουν μόνο με το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και τη ροή ε, κεφαλαίων, αλλά είναι και στενά συνειφασμένα θέματα με την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Και τώρα ξαναδίνω το λόγο στους ομιλητές μας, αν το επιθυμούν, για να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ. Θα είμαι συντομότατος. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου. Με την ε, ανάδειξη Τραμπ από την πρώτη μέρα δηλαδή, δεν πρόλαβε να γίνει πρόεδρος, απέσυρε την υπογραφή του από τη συμφωνία TAPP. Μετά ο Πρωθυπουργό Άμπε προσπάθησε συνέπεια να πείσει τον κύριο Τραμπ να αποδεχθεί την αξία της TAPP περίπου 40% του παγκοσμίου ΑΕΠ καλύπτεται από εκεί. Επίσης, αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι πρόκειται για μια συμφωνία όπως η ΣΕΤΑ με τον Καναδά και την Ευρώπη. Δεν πρόκειται για ρυθμίσεις μηδενικών δασμών μόνο. Η TPP ε, εισήγαγε υψηλά πρότυπα για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ε, προστασίας των επενδύσεων, ε, προστασίας διανοητικών δικαιωμάτων, τέτοιες διασφαλίσεις. Το Κοινοβούλιο θέλει να διασφαλίσει ψηλά πρότυπα περιβαλλοντικής προστασίας, εργατικών, εργασιακών δικαιωμάτων κλπ. Όλα αυτά ενσωματώνονται στην ε, TPP. Θα ήταν μεγάλη απώλεια αν δεν τεθεί σε ισχύ η συμφωνία TPP. Πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Αν δεν επιστρέψουν οι ΙΠΑ στην TPP με την παρούσα δομή της, δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ η TPP. Μεταξύ των 11 συμβαλωμένων χωρών, η ε, Χιλή, η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία, η Ιαπωνία βέβαια. Ε, γίνονται συζητήσεις, γίνονται συζητήσεις μεταξύ των συμβαλωμένων σχετικά με το τι πρέπει να γίνει στο μέλλον. Κάποιοι λένε γιατί να μην συμφωνήσουμε οι 11 και μετά να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Άλλοι λένε, αν δεν έρθουν οι ΙΠΑ, γιατί να μην καλέσουμε να έρθει η Κίνα ή η Κορέα. Δεν νομίζω όμως ότι η Κίνα θα προσχωρήσει στην TPP. Τώρα πιέζουν ε, υπέρ μιας ε, περιφερειακής συμφωνίας, ε, η 10 ΑΣΕΑΝ, η Ινδία, η Νέα Ζηλανδία και η Κίνα. 16 συνολικά. Αυτό είναι κάλυψη εντυπωσιακή. Δηλαδή είναι μεγάλο το ΑΕΠ που καλύπτει μια τέτοια συμφωνία. Ε, εμείς α, είχαμε και το ΕΦΤΑΠ, Συμφωνία Ελευθερών Συναλλαγών στην ε, περιοχή του Ειρηνικού και της Ασίας και εκεί καλύπτονται 18 χώρες. Τώρα η διακυβέρνηση Τραμπ θέλει διμερείς και όχι πολυμερείς συμφωνίες. Προς το παρόν η Ιαπωνία συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη μιας καλής συμφωνίας στα πλαίσια του Άρσεπ. Αλλά βέβαια δεν θέλω να επικρίνω κανέναν, αλλά σε, αυτή, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και συμφωνίες πάντα κάποιες χώρες θέλουν πολύ να έχουν μια συμφωνία σε χαμηλό επίπεδο ποιοτικά και το θέμα είναι πρέπει να το δεχτούμε αυτό. Νομίζω όχι. Αν λοιπόν άλλοι εταίροι επιθυμούν να ε, υπογράψουν μια συμφωνία για την ΑΡΣΕΠ θα ζητήσουμε να είναι σε υψηλότερο επίπεδο ποιοτικό αυτή η περιφερειακή συμφωνία. Και η Κίνα και η Ινδία φαίνονται πολύ απρόθυμες. Λένε γιατί να μην κάνουμε τώρα συμφωνία άμεσα. Εμείς λέμε όχι. Θέλουμε να διαπραγματευτούμε και να μιλήσουμε περισσότερο ο Πρωθυπουργός ε, συνέχισε να συνομιλεί με τον κύριο Τραμπ για να τον πείσει για τα υπέρ μιας πολυμερούς συμφωνίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι θα κάνει κάτι παρόμοιο. Γιατί εδώ χρειάζεται συνεργασία μεταξύ μας, η Ιαπωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να πείσουμε τις Ηνωμένε Πολιτείε να επανέλθουν στη συμφωνία. Αυτή είναι η στρατηγική μας. Ευχαριστώ. Διευθυντά Βίγκαν, θέλετε να πείτε κάτι. Ευχαριστώ ο, η Επίτροπος για το Εμπόριο και οι συνάδελφοι από το, υπεύθυνοι για το εμπόριο έχουν δώσει απαντήσεις ε, στο Κοινοβούλιο για αυτά τα θέματα. Εγώ τονίζω ότι συμφωνούμε πάρα πολύ με την ανάλυση που έκανε ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας. Παρόλο που δεν είμαστε μέρη στη συμφωνία αυτή, ε, λυπούμεθα που δεν δόθηκε συνέχεια στη συμφωνία TPP από την Αμερικανική κυβέρνηση. Δεν πρόκειται μόνο για δεσμεύσεις πρόσβασης στην αγορά, αλλά και για την ε, θεσμοθέτηση προτύπων σε μια ευρύτατη περιφέρεια που συμπεριλαμβάνει ε, τον Ειρηνικό και χώρες από την Ασία και τη Λατινική Αμερική. Δηλαδή ήταν μια καλή συμβολή στο πολυμερές εμπόριο Στου κανόνε για επενδύσει και πρότυπα σε πολλού άλλου τομεί. Ήταν μια συμφωνία θεσμοθέτηση προτύπων. Αυτό είναι κάτι που ενδιαφέρει ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που κάνει στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξει ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο παντού. Έτσι θα είναι και θεμητή μια παρόμοια συμφωνία αν έχουμε υψηλά πρότυπα και κοινωνικά και ε, περιβαλλοντικά, πρότυπα προϊόντων, ε, εργασίας κλπ. Και εδώ υπάρχουν διάφορες επιλογές για τα συμβαλόμενα μέρη. Ακόμα δεν έχει λεχθεί η τελευταία λέξη. Ε, πριν από λίγες μέρες είχαν γίνει συζητήσεις άλλη μια φορά. Ένα είναι σαφές, δεν μπορεί να υποκαταστήσει η Κίνα τις Ηνωμένε Πολιτείες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν απλουστευτικό κάτι τέτοιο. Ε, υπάρχουν ε, πολλές δεσμεύσεις που έχουν να κάνουν με την τεράστια αμερικανική αγορά. Οι εναπομένουσες χώρες, οι εναπομείνωσες χώρες μπορούν βέβαια να επικυρώσουν τη συμφωνία αυτές. Και το, η προϋπόθεση του ε, ΑΕΠ των δύο τρίτων φαίνεται ρεαλιστικό αφού αποσύρθηκαν οι ΙΠΑ. Αλλά Αυτές είναι αποφάσεις που δεν θα λάβουμε εμείς. Ε, την ανάλυση του πρέσβη εις ό,τι αφορά την συνεργασία, τη συμφωνία συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτή είναι μια πιο επίπεδη συμφωνία βέβαια, η οποία δεν πληρεί τις ίδιες προϋποθέσεις, ούτε θέτει πρότυπα με το σωστό τρόπο. Βέβαια, ε, ένα πράγμα πρέπει να τονίσουμε σε αυτή τη συζήτηση ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενθαρρυντικό να προωθήσει τη δική της ε, πολιτική που προάγει το εμπόριο στην περιοχή. Στη Σιγκαπούρη την ε, τελευταία εβδομάδα ε, πριν από τη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών Ασιαν και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, συζητήθηκε το θέμα αυτό. Έχουμε 11 συμφωνίες, ε, δηλαδή δυνητικές συμφωνίες και η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Άμπε ήταν πολύ θετική. Εμείς φέτος θέλουμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα και εις ό,τι αφορά τη νέα στρατηγική συμφωνία με την Ιαπωνία και για συμφωνία ελευθερών συναλλαγών. Ε, έχουμε με την Κορέα μια τέτοια συμφωνία, έχουμε οριστικοποιήσει τις διαπραγματεύσεις με την Κορέα και το Βιετνάμ, γίνονται με τις Φιλιππίνες διαπραγματεύσεις όπως και με την Ινδονησία, ε, έχουμε διαπραγματεύσεις με την Κίνα και την Ινδία για... Ο, η, ε, με την Ινδία έχουμε ελευθέρων συναλλαγών, ε, αλλά οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές. Δηλαδή υπάρχει εμπορική πολιτική πολύ δυναμική από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ζήτηση είναι σημαντική και οι Υπουργοί Οικονομικών αποφάσισαν ότι θα πρέπει να δούμε και αν υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν συμφωνίε ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ περιφερειών. Μπορώ παρακαλώ να ρωτήσω κάτι πολύ σύντομα. Η συμφωνία της Σικαπούρης Ισχύει γιατί αναφερθήκατε. Ναι. Και σίγουρα θα ολοκληρωθεί σύντομα. Στο μέλλον όμως θα έχουμε την απόφαση. Οπότε τότε θα ξέρουμε περισσότερα. Πρόεδρος, ναι, είναι πολύ σημαντικό για τα θέματα της αρμοδιότητας. Παρακαλώ κυρία Φαλών. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούσαμε πολλά καλά σχόλια από τους δύο προλαλήσαντες. Εγώ θέλω να προσθέσω το εξής. Όταν ήταν ε, εδώ στις Βρυξέλλες ο σύμβουλος του Πρόεδρου της Κίνας είχε πει ότι θα ήταν πολύ καλό το Δηλαδή αντιλαμβάνονται την ε, μεγάλη στρατηγική σημασία που έχει η συμφωνία και βέβαια μετά τόσα είπε ο πρόεδρος Τραμπ, δεν τους ευχαριστεί. Ελπίζω πάντως ο Πρωθυπουργός Άμπε της Ιαπωνίας να πείσει για να δοθεί συνέχεια στο TTIP. Η προσέγγιση του Τραμπ δεν λειτουργεί. Είναι εντελώ διαφορετικό το να είσαι επιχειρηματίας και εντελώ διαφορετικό να κάνεις διεθνή πολιτική. Ο Πρωθυπουργό Σάμπε συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και έκανε τις διαπραγματεύσεις για έξι χρόνια. Θα είναι μεγάλη η οικονομική και πολιτική απώλεια. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, κυρίες και κύριοι εκ μέρους των Ευρωβουλευτών μας που συμμετείχαν στην συζήτηση αυτή. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους τους προσκεκλημένους μας που ήρθατε σήμερα. Την κυρία Φαλόν, ετοιμαζόμαστε, όπως ξέρετε, για την αποστολή μας στην Ιαπωνία. Και σήμερα το απόγευμα θα συνεχίσουμε να συζητάμε για την περιοχή. Έτσι μπορούμε να συνεισφέρουμε στη συζήτηση που γίνεται για την ασφάλεια στην περιοχή. Θα μιλήσουμε δηλαδή για την ε, Νότια Συνική Θάλασσα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και ένα θερμό χειροκρότημα για όλους σας. Μικρή διακοπή, παρακαλώ, για να αλλάξουν οι ομιλητές εδώ στο βήμα.